έχουν εγκριθεί. Τους τίτλους λοιπόν μπορείτε να του βρείτε στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής. Και τώρα κυρίε και κύριοι, σα παρακαλώ να λάβετε υπόψη τι εξή αποφάσει. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στι 11 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το άρθρο 146.3 του κανονισμού η σύνοδο της 8 και 9 Οκτωβρίου να διαγραφεί προκειμένου να υπάρχει απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία της ε, ψήφου για το σώμα των επιτρόπων που θα λάβει, η θα λάβει χώρα 20 με 23 Οκτωβρίου. Άρα 8 και 9 Οκτωβρίου ε, η σύνοδο τη Βρυξέλλα που προβλεπόταν καταπίπτει. Αυτά λοιπόν ως προς τις ανακοινώσεις μου κυρίες και κύριοι και τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Σύμφωνα με τον άρθρο 149 εγκρίθηκε λοιπόν